Παρακαλώ κυρίες και κύριοι, καθίστε στις θέσεις σας για να μπορέσουμε να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Πρώτα απ' όλα καλωσορίζω εδώ θερμά τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Χαιρετίζω φυσικά και τους συναδέρφους μου ευρωβουλευτές. Και όλος ιδιαίτερος χαιρετίζω εδώ τον κύριο Σορίν Λαζάρ, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, Δημοσιονομικών και Τραπεζών του Κοινοβουλίου της Ρουμανίας, ο οποίος ε, θα καταλήξει και σε συμπεράσματα στο τέλος της συνάντησης αυτής όσον αφορά τις προτεραιότητες επενδύσεων μετά το 2020 για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα επικεντρωθούμε εδώ στην προτεραιότητα των επενδύσεων. Παρά τις διάφορες πρωτοβουλίες για να διορθωθεί η κατάσταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρει ακόμα από σημαντική έλλειψη επενδύσεων. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο πρόγραμμα, το Invest EU, ακριβώς για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Η πρόταση αυτή της Επιτροπής βασίζεται στην επιτυχία των Ευρωπαϊκών Ταμείων Στρατηγικών Επενδύσεων. Το πρώτο ταμείο και το δεύτερο ταμείο. Το πρώτο ξεκίνησε το 2015 και το δεύτερο το 2018. Πρόκειται για δύο ταμεία τα οποία έδωσαν την απαραίτητη όθηση στις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως πρέπει να πάμε ακόμα πιο μακριά, κυρίως για να στηρίξουμε υποδομές βιώσιμες, την έρευνα, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις κοινωνικές επίσης επενδύσεις και υποδομές. Δρώντας λοιπόν γρήγορα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Έτσι στις 16 Ιανουαρίου Τώρα, στι αρχέ της χρονιάς ενέκρινε εντολή διαπραγματεύσεων το Κοινοβούλιο με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε το πρόγραμμα InvestEU που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκριθεί οριστικά. Υπήρξαν τροπολογίες οι οποίες αυξάνουν μεταξύ άλλων την εγγύηση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι 40,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές για κινητοποίηση παραπάνω από 698 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε εγγύηση για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 38 δισεκατομμυρίων ευρώ για να κινητοποίησε 650 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν, τώρα πια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να μπει σε διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς, με το Συμβούλιο δηλαδή, υπό την Ρουμανική Προεδρία βέβαια. Πριν ολοκληρώσω, πρέπει να σας πω ότι πρέπει να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, ώστε την 1η Ιανουαρίου του 2021 να είναι όλα έτοιμα και το πρόγραμμα να μπορέσει να υλοποιηθεί αμέσως τότε έχετε μπροστά σας και κάποιες κάρτες που μπορείτε να συμπληρώσετε εάν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις. Ξέρετε πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, το έχετε ήδη χρησιμοποιήσει και χτες και σήμερα το πρωί. Αν θέλετε λοιπόν το λόγο, παρακαλώ να συμπληρώσετε αυτές ε, τις καρτούλες που έχετε μπροστά σας και μετά από τις αρχικές παρουσιάσεις θα δώσω το λόγο διαδοχικά σε δύο ε, βουλευτές οι γερουσιαστές από τα Εθνικά Κοινοβούλια και στη συνέχεια σε έναν Ευρωβουλευτή και ούτω καθεξής. Όπως και εσείς και εγώ λυπάμαι που δεν είναι εδώ ο κύριος Ζέρκη Κατάινεν που είναι Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λυπάμαι που δεν μπορεί να είναι μαζί μας στις Βρυξέλλες σήμερα και ούτε κανένας άλλος επίτροπος δεν μπόρεσε να τον αντικαταστήσει σήμερα το απόγευμα. Οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Βέρνερ Χόιερ που είναι ο πρόεδρος της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και θα πάρει το λόγο για το πολύ πέντε λεπτά. Παρακαλώ πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πραγματικά είναι δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσω, να καταφέρω. Κύριε και κύριοι, με μεγάλη χαρά ήρθα εδώ να σας μιλήσω σήμερα στις Βρυξέλλες και να σας μιλήσω για ένα από τα θέματα κλειδί που θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, είναι, όχι απλώς ενδιαφέρεται, αλλά είναι και για αυτή είναι ένα καυτό θέμα, το θέμα των επενδύσεων. Και εκείνη δημιούργησε και προσπάθησε να πείσει και τους άλλους για το σχέδιο Juncker, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Πρόκειται για πολύ θαραλέα μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν στην εποχή τους και ευχαριστώ πάρα πολύ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα νομοθετικά σώματα που πήραν αυτή τη θαραλέα απόφαση. Γιατί το να βγάζουμε χρήματα από τις επιδοτήσεις και να τα βάζουμε σε μια διευκόλυνση εγγύσεων δεν είναι μια εύκολη απόφαση για κανέναν. Ε, την πήρατε όμως και πετύχαμε. Τώρα το Invest EU προχωράει προς μια αντίστοιχη κατεύθυνση. Ο βασικό κανόνα λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να είναι να δούμε τι λειτουργήσε καλά, ας το κρατήσουμε και α αλλάξουμε και α βελτιώσουμε ότι δεν λειτουργήσε αρκετά καλά ή θα μπορούσε να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Δηλαδή με δύο λόγια πρόκειται για μια σαφή επιτυχία. Σήμερα οι επενδύσει καθορίζουν το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κοινωνιών τη. γιατί έχουν ε, επίδραση για πολλές δεκαετίες μετά. Τι θέλουμε λοιπόν να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια και πού βρισκόμαστε σήμερα. Μια αιτία για την άνηση και αργή ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει να κάνει με την κρίση στην οποία μπήκαμε πριν από μία δεκαετία. Αν βέβαια σκάψουμε λίγο πιο βαθιά θα διαπιστώσουμε ότι η ανάκαμψη και τα επίπεδα ανάπτυξης εξακολουθούν να διέπονται από κάποιε διορθωτικέ αδυναμίες. Πρώτα απ' όλα η Ευρωζώνη εξαρτάται κατά πολύ ε, στην ε, στήριξη των πολιτικών. Και υπάρχουν πολλά στοιχεία που εξακολουθούν να είναι ευάλωτα. Οι αγορές εξαρτώνται από την χρηματοδότηση και δεν υπάρχει αρκετή ολοκλήρωση στη χρηματοδότηση κεφαλαίων και μηχανισμών χρηματοδότηση. Έπειτα υπάρχει άνηση ανάπτυξη ανάμεσα σε περιφέρειε και σε χώρε. Αντί να αναπτυσσόμεθα όλοι λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο μαζί, εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλήσει και μεταξύ αλλά και μέσα σε μία και την ίδια χώρα μέλο. Οπότε η Ευρώπη δεν πετυχαίνει το στόχο τη της συντοχή. Έπειτα, υποφέρει η Ευρώπη από το γεγονό ότι μειώνεται η ανταγωνιστικότητα, αν τη συγκρίνουμε με την Βόρεια Αμερική και την Ασία και το χάσμα που ξεκίνησε στις αρχές του 2000 μεγαλώνει. Κάτι το οποίο είναι μια ανησυχητική τάση για πολλούς λόγους. Επίσης μειώνεται ο πληθυσμός στην Ευρώπη. Η γύρανση του πληθυσμού αυξάνεται. Η παραγωγικότητα μόνο όταν είναι πάνω από το μέσο όρο θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Η ανάκαμψη επίσης των επενδύσεων είναι ανεπαρκής. Στον ιδιωτικό τομέα κυρίως δεν είναι αρκετές ούτε υπάρχουν αρκετές επενδύσεις στις υποδομές, στην ε, εκπαίδευση, στην ε, καινοτομία και την έρευνα. Χρειάζονται επίσης ισορροπημένοι προπολογισμοί. Τα δημοσιονομικά μειώθηκαν κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κρίση. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα δούμε μαζί όλους αυτούς τους παράγοντες, δείχνουν ότι χρειάζονται διαρθρωτικές ε, αλλαγέ για την σύγκληση, για την βελτίωση των συνθήκων ζωής. Πρέπει να επικεντρωθούμε στις επενδύσεις, αντιμετωπίζοντας τις ε, αδυναμίες, για να είμαστε πιο ανθεκτικοί στο μέλλον. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αυτό ακριβώς κάνει. Είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 60 χρόνια που λειτουργεί αυτή, οι χώρε ε, μέλη έχουν πληρώσει 40 δισεκατομμύρια μόνο για τις ε, μετοχές ε, της τράπεζας. Και τα ποσά αυτά μας βοήθησαν στα 60 χρόνια πάνω από 1,13 να επενδυθούν που οδήγησαν σε πάνω από 3-3 Συνεπώ, τα χρήματά μα πιάνουν τόπο. Όχι το φορολογούμενο, αλλά τα χρήματα τα οποία εμεί συγκεντρώνουμε από επενδύσει. Και έτσι έχει βελτιωθεί η ζωή των Ευρωπαίων όλα αυτά τα χρόνια. Χρειάζονται όμω και άλλε προσπάθειε και αυτό ξεκίνησε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Χτίζουμε λοιπόν πάνω σε αυτέ τι επιτυχίε. Κυρίε και κύριοι, αν έχουμε τη φιλοδοξία να πετύχουμε του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ και του στόχου για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή των Παρισιών πρέπει να κινητοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα. Τα χρήματα των φορολογούμενων δεν πρόκειται να φτάνουν για να πετύχουμε του στόχου αυτού. Το InvestEU λοιπόν, κατά τη γνώμη μα, τροποποιεί το ΕΦΣΥ και το καταστά ένα μακροχρόνιο μηχανισμό για να στηρίσει επενδύσεις στον τομέα της ε, σύγκλησης, της καταπολέμησης, κλιματικής αλλαγής κλπ. Κυρίες και κύριοι, για 15 χρόνια συνεχώς εμείς βρισκόμαστε πίσω από τους ανταγωνιστές μας στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Κίνα με το 1,5% του ΕΠΑ. 1,5% 15 χρόνια τώρα, κάθε χρόνο λιγότερο από αυτούς. Κάτι το οποίο οδηγεί σε μείωση της ανταγωνιστικότητάς μας και της ανάπτυξης της παραγωγικότητάς μας. Αυτό ακριβώς πρέπει να αλλάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Ανεμή Τόρτεμπούμ, μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Το οποίο Ελεκτικό Συνέδριο ασχολήθηκε με το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και έχει καταλήξει σε ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις για την ολοκλήρωση της λειτουργίας αυτού του ταμείου. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ως ελεγκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ρόλος μου είναι να εστιάσω το ενδιαφέρον μου στον τρόπο με τον οποίο ξοδεύεται το ευρωπαϊκό χρήμα. Δεν αφισβητούμε τι πολιτικέ προτεραιότητε για την επενδυτική στήριξη αυτέ Εξετάζουμε πόσο καλά χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα υφιστάμενα εργαλεία για να διοχετεύσει κονδύλια να εξυπηρετήσουν τις ε, πολιτικές προτεραιότητες. Και αυτό είναι κάτι που έχει αλλάξει με τα πρόσφατα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια. Έχουμε το EFSI και το InvestEU, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και το Ταμείο InvestEU, EU, επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Και κάθε, όπως κάθε παραδοσιακό σύστημα ενίσχυσης πρέπει να γίνονται αντικείμενο χρηστής διαχείρισης και να εξετάζονται από τα κοινοβούλια. Αυτό είναι και ο ρόλο μα. Να αξιοποιήσουμε του ελέγχου για να βοηθήσουμε τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσουν κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εκτό από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και το νέο πρόγραμμα InvestEU Επενδύστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικό, βασική πηγή ευρωπαϊκή στήριξη για τι επενδύσει το 2021 με 2017. 21 με 27 μάλλον. Θα λειτουργήσει με μια εγγύηση 38 εκατομμυρίων ευρώ από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αύξηση κατά 26 ε, ε, ευρώ εγγύηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο στρατηγικών επενδύσεων. Το InvestEU λοιπόν θα χτίσει πάνω στην εμπειρία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και θα αντικαταστήσει και διάφορα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι μια απλούστευση ευπρόσδεκτη σε σύγκριση με τι τρέχουσε υφιστάμενε ρυθμίσει. Το InvestEU θα λειτουργεί πάνω στι ίδιε γραμμέ όπω το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, παρόλο που μπορεί να υπάρξουν διαφορέ στη διακυβέρνηση. Το Ελεκτικό Συνέδριο δημοσίευσε μια έκθεση για την λειτουργία των πρώτων τριών ετών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών στρατηγικών επενδύσεων, 1,0. Συμπεραίνουμε ότι ήταν επιτυχημένη η λειτουργία αυτού του Ταμείου του Στρατηγικού για τις επενδύσεις, αλλά παραμένουν προκλήσεις για να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία το εγχείρημα αυτό. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλιά μας έχουν να κάνουν με τις μελλοντικέ δράσεις του InvestEU και θέλω να σταθώ σε αυτά τα σχόλιά μας στην έκθεσή μας για να αναδείξω πέντε βασικές προκλήσεις. Η πρώτη πρόκληση είναι να προσαρμόσουμε τις χρηματο... τα χρηματοπιστωτικά και χρηματοδοτικά προϊόντα στις ανάγκες. Βάσει του Ταμείου Στατικών Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, ανέλαβε χρηματοδότηση υψηλότερου ρίσκου ε, προσφέροντας επενδυτικά δάνεια κατηγορίας senior, τα κλασικά, με μεγαλύτερη και πιο μακροχρόνια περίοδο λήξης και έχοντας, υιοθετώντας επισφαλείς θέσεις, μη καλυμμένες θέσεις, όταν είχε να κάνει με ομολόγους της υψηλού κινδύνου σχετικά ε, μικρή χρήση έγινε άλλων ε, χρηματοπιστωτικών προϊόντων διαθέσιμων υψηλού κινδύνου. Εμείς ε, συστήνουμε η Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων να προωθήσει τη χρήση προϊόντων υψηλότερου κινδύνου μόνο σε τεκμηριωμένες περιπτώσεις για να διασφαλίσει ότι η επενδυτική στήριξη λειτουργεί συμπληρωματικά σε αυτή που παρέχουν οι εθνικές τράπεζες οι επενδυτικές για την προώθηση και θα στοχευτούν καλύτερα τα κενά της αγοράς. Δεύτερη πρόκληση είναι να αποφύγουμε τον ανταγωνισμό με άλλε πηγέ κοινοτικών κονδυλίων. Το ΕΦΣΥ εν μέρει αντικατέστησε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία στου τομεί των μεταφορών και τη ενέργεια και ε, τονίζουμε το ότι μπορεί να υπάρχουν επικαλύψει μεταξύ του ΕΦΣΥ, του στρατηγικών επενδύσεων δηλαδή, και των λοιπόν διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Προτείνουμε η Κομισιόν να υιοθετήσει μέτρα για να ενθαρρύνει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των εργαλείων και να αποφευθεί ο ανταγωνισμό μεταξύ αυτός. Η πρόταση, αυτών. Η πρόταση για το InvestEU για μία και μόνη εγγύηση του προπολογισμού που θα αντικαθιστά τα υφιστάμενα, πολλέ εγγύησει για τα υφιστάμενα ε, εργαλεία, πηγαίνει προ τη σωστή κατεύθυνση. Η τρίτη πρόκληση είναι να διασφαλίσουμε την προσθετικότητα των project που στηρίζουμε. Δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι τα νέα project θα έχουν χρηματοδότηση και θα υπάρχουν που δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και να υλοποιηθούν χωρί την ευρωπαϊκή στήριξη. Στον έλεγχό μα, το ΕΦΣΥ είδαμε ότι ορισμένα project θα μπορούσαν να έχουν γίνει χωρί στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Συστήνουμε να ενισχυθεί η αξιολόγηση του κατά πόσο η στήριξη από αυτό το ταμείο μπορεί να αντικαταστήσει άλλε πηγέ χρηματοδότηση. Τέταρτη πρόκληση είναι να κάνουμε ισχυρέ εκτιμήσει τη επένδυση που ουσιαστικά κινητοποιείται. Είναι δύσκολο να δούμε κατά πόσο ευρωπαϊκή στήριξη παίζει αποφασίσει αποφασιστικό ρόλο στο να προχωρήσει και να καρποφορήσει μια νέα επένδυση, γιατί εμπλέκονται εκεί και άλλε πηγέ χρηματοδότηση, δημόσιε και ιδιωτικέ. Ε, στην έκθεσή μα, λοιπόν τονίζουμε ορισμένε περιπτώσει, όπου θεωρούμε ότι οι επενδύσει που κινητοποιήθηκαν υπερέβησαν το ποσό των ε, επιπρόσθετων επενδύσεων που θα μπορούσαν να είχαν αποδοθεί λογικά στη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών επενδύσεων. Συστήνουμε λοιπόν να βελτιωθεί η μεθοδολογία για την αξιολόγηση αυτή. Και τέλος, πέμπτη πρόκληση είναι να επιτύχουμε σωστή απορρόφηση της στήριξης. Έχουν εκφραστεί ανησυχίες στα κράτη-μέλη για τη γεωγραφική κατανομή τη στήριξη τη επενδυτική που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τουλάχιστον τα πρώτα τρία χρόνια τη λειτουργία του. Σημειώνουμε ότι 15 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση με καλά εδρεωμένε εθνικέ επενδυτικέ τράπεζε, αυτέ οι χώρε είναι που το αξιοποίησαν περισσότερο. Άρα δείχνει αυτό ότι η ικανότητα των κρατών μελών να δημιουργούν project και έργα υψηλή ποιότητα είναι καθοριστικό παράγοντα για τον το πού θα καταλήξει η επενδυτική στήριξη και ποιος τελικά θα την χαρεί. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκαν τις συστάσεις μας να εξετάσουν τις ε, βασικές δομικές αιτίες πίσω από την κατανομή τη στήριξη που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτή η μελέτη θα είναι χρήσιμη για την υλοποίηση του προγράμματο Invest EU. Και αν υπάρχουν ζητήματα στην πλευρά τη προσφορά, τότε ο ρόλο του Συμβούλου και τη τεχνική βοήθεια είναι ακριβώ εξαιρετικά σημαντικό και για το επόμενο πρόγραμμα, το Invest EU. Κύριε Πρόεδρε, με αυτά τα συμπεράσματα μπορεί κανείς να έχει μια άποψη για τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ε, πλευρά του ελεγκτικού ε, συναδρίου και για το ποια είναι η άποψή μας για όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το InvestEU μπορεί να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ε, βελτιώσουν το έργο τους και να ε, σταθούν στο ύψος των προκλήσεων ε, που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ πράγματι είναι επιτυχία το Ευρωπαϊκό Ταραμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θέλω να δώσω το λόγο στον Χωσέ Μανουέλ Φερναντέ, έναν από τους προτεργάτες του κειμένου που ήταν συνεισηγητής για το θέμα αυτό. Κύριε Φερναντές, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συνεχίσω με το Invest EU και θα ήθελα να μιλήσω στα πορτογαλικά, αν μου επιτρέπετε. Στην πρότασή μας, η οποία υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, δεν γίνεται λόγος για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξού και επειδή υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, γίνεται λόγος για την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέλουμε να ανεβάσουμε τα εγγυημένα ποσά να ξεπεράσουν το 40, κάτι δις ευρώ, διότι θέλουμε να διατηρήσουμε το ύψος των εγγυήσεων για τα τρία άλλα κοινοτικά ε, χρηματοδοτικά εργαλεία. Από το 2021 μέχρι το 2027 δεν έχει κανένα νόημα να μειώσουμε τις εγγυήσεις των χρηματοδοτικών εργαλείων. Δεν Πρόκειται για παράταση του σχεδίου Juncker του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Είναι το ΕΦΣΥ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, συν τα άλλα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχουμε τι υποδομέ, την έρευνα, την καινοτομία, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και τον κοινωνικό πυλώνα. Αυτά είναι τα πεδία που μα απασχολούν και θέλουμε να ενισχύσουμε τον κοινωνικό πυλώνα και να ενισχύσουμε τη στήριξη που δίνουμε στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Το Invest EU, λοιπόν, το επενδύστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υφίσταται. Είναι ένα ανοιχτό ταμείο το οποίο ε, θα συνδέεται με αυτούς που προγραμματίζουν τη διαχείριση των κονδυλίων. Αυτή είναι νέα απέτηση και για τις περιφέρειες αλλά και για τις πληρωμές. Δηλαδή, δεν είναι σκοπός μας να αντικαταστήσουμε την πολιτική συνοχή με αυτό το εργαλείο καθόλου, τον αντίον. Η υποχρέωσή μας είναι να συμπληρώσουμε την πολιτική συνοχή και να υπάρχουν συνέργειες και η ύπαρξη συνεργειών είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Θεωρώ ότι το πιο θεμελιώδες που παρουσιάζει η πρότασή μας είναι η ενίσχυση της πλατφόρμας συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται στους επενδυτές. Είναι κεφαλαιόδου σημασία κάθε κράτος μέλος, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε περιφερειακό επίπεδο, να κάνει τη δουλειά που του αναλογεί και να διαθέτει αυτή τη πλατφόρμα συμβουλευτικής στήριξης στους επενδυτές για να βρεθούν νέες λύσεις, για να βρουν στέγη, τα μικρά έργα και τα νέα έργα και για να ε, κινηθούν αυτές οι επενδυτικές πλατφόρμες. Ελπίζω πράγματι να καταφέρουμε να φτάσουμε σε απλούστευση. Ξέρετε, συχνά όταν η Επιτροπή λέει ότι απλουστεύει τα πράγματα, αυτό πιο μάλλον ανησυχητικό ακούγεται παρά θετικό. Ελπίζω όμως να διαψευστώ αυτή τη φορά να ισχύσει και να υπάρχει αληθινή απλούστευση. Η γεωγραφική ε, ισορροπία είναι εξίσου σημαντικό στοιχείο, όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το είδος της δραστηριότητας. Επιμένω σε αυτή την πλατφόρμα συμβουλευτικής στήριξη σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Κάτι το καινούργιο στο InvestEU είναι το εξή και πρόκειται περί καινοτομίας. Το σύνολο της εγγύησης δεν θα κατευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Τραπεζα Επενδύσεων. Θα έχουμε 25% για τα εθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ε, τα επενδυτικά. Και αυτό γύρει νέε προκλήσεις για τα κράτη-μέλη, τα οποία πρέπει να θεσπίσουν αυτές τις ε, επενδυτικές τράπεζες ή τις αναπτυξιακές, να ενισχύσουν τις ήδη υφιστάμενες, να ανοίξουν έτσι ώστε να λειτουργήσουν αυτού του είδους τα τραπεζικά σχήματα σε χώρες που δεν υπάρχουν. Κάτι το σημαντικό για τα κράτη-μέλη που δεν έχουν τέτοιου είδους ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι το εξής. Πέρα από την ενίσχυση των εγγυήσεων, πέρα από το ύψος αυτού του ποσού της εγγύησης, τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν ένα μέρος του χρηματοδοτικού φακέλου για ε, συγκεκριμένα έργα. Δηλαδή, ένα μέρος του εθνικού φακέλου μπορεί να αντικατασταθεί από διαρθρωτικά ταμεία και να μπει στο InvestEU. Δηλαδή κινητοποιούνται πόροι που έχουν βαθμολόγηση τριπλού α και έτσι αποφεύγουμε το σκόπελο των κρατικών ενισχύσεων. Αυτό είναι καλό νέο για τα κράτη-μέλη, τα οποία συνάπτουν εταιρικέ σχέσεις και κατά τη σύναψη αυτών των συμφωνιών μπορούν να αφρίσουν το κονδύλια του Ταμείου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, του Ταμείου Συνοχής με τα κονδύλια και τα εργαλεία των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και διαθέτουν ε, μια πλειάδα εργαλείων δηλαδή ε, για να ε, προχωρήσουν τα έργα. Μιλήσαμε για την προσθετικότητα, για το αθρηστικό αν θέλετε αποτέλεσμα. Στο InvestEU δεν βάζουμε τον ίδιο ορισμό όπως αυτό που βάλαμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Γιατί η προσθετικότητα για ένα κοινωνικό πρόγραμμα δεν είναι ίδια με την προσθετικότητα ενός έργου που έχει σαν στόχο τη δημιουργία υποδομών. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την πρότασή μας γιατί εισάγει και βελτιώνει τη διαχείριση. Γιατί δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους και αναφέρομαι εδώ στις περιφερειακές επενδυτικές τράπεζες για παράδειγμα και στην Επιτροπή των Περιφερειών και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα λοιπόν σε όλους αυτούς να διαδραματίσουν ένα ρόλο πιο πρωταγωνιστικό, πιο ενισχυμένο. Η πρότασή μας εδράζεται σε στέρεες βάσεις και ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα κάνει ε, τη δουλειά που του αναλογεί. Ξέρετε, ε, ακούσαμε ότι ίσως το Φεβρουάριο θα υπάρξει εντολή διαπραγματεύσεων με εμάς το περιμένουμε. Αλλά επειδή περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειμονούμε λίγο. Δεν θα περιμένουμε επάπειρον και επαόριστον, ούτε εμεί ούτε η Ευρώπη. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πραγματικά δώσει αυτόν τον αγώνα από την αρχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ο κύριος Τζούλιαν Γιανκουτόρα, πρόεδρος της Υπηρεσίας Βιομηχανίας του Κοινοβούλιο της Ρουμανίας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω προετοιμάσει πέντε διαφάνειες. Μου είπαν ότι δεν γίνεται όμως να τις δείξω. Οπότε θα μιλήσω στην μητρική μου γλώσσα. Οπότε. Κοιτάξτε, ε, φτάνουμε στο τέλος της συζήτησής μας εδώ στο Κοινοβούλιο και ακριβώς Θέλουμε να καταλήξουμε σε κάτι που να μπορεί να ισχύει σε όλες τις χώρες μέλη, ουδέτερο, χωρίς ε, διακρίσεις σε βάρος κανενός και λαμβάνοντας υπόψη μας όλους τους παράγοντες, τους μακροοικονομικούς, τους προπολογισμού, τις χώρες μέλη και την Ευρωζώνη. Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για το σύμφωνο σταθερότητας, μιλάμε για πολιετή προπολογισμό και για την ανάγκη να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους, όπως είναι η σύγκληση, η ανταγωνιστικότητα, το ανθρώπινο κεφάλαιο, επενδύσεις, επενδύσεις στην έρευνα, στην ανάπτυξη και την κοινοτομία. Επίσης, χρειάζεται σύγκληση και συνοχή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, ποια είναι η πραγματικότητα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχουν μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες δεν εξηγούνται πάντα Υπάρχουν ελλείμματα στους τρέχοντες λογαριασμούς. Υπάρχουν οικονομικές φούσκες, οι οποίες ε, δεν ε, μπορεί να συνεχίζονται και σαφώς και χρειάζονται επενδύσεις. Αυτή είναι μια πεποίθηση την οποία συμμεριζόμαστε όλοι. Ποιε είναι αυτές οι επενδύσεις λοιπόν οι αναγκαίες που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις αναλύσεις που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που δείχνουν ότι σταθερότητα τιμών είναι αναγκαία. Σταθερότητα τιμών. Επαναλαμβάνω. Δεύτερον, ενιαία αγορά. Και τρίτον, τιμές και ικανότητα παραγωγής έτσι ώστε όλοι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι, ποια θα ήταν αυτή η θαυματουργή λύση για να την κατανοήσουμε καλύτερα θα σας δώσω κάποια νούμερα. Πληρώνουμε 1,13 δισεκατομμύρια την ημέρα για την ενέργειά μας, σε λογαριασμούς για την ενέργεια. Ό,τι πιο ακριβό υπάρχει στον κόσμο. Δεύτερον, ο λογαριασμός αυτός πλήττει την ανταγωνιστικότητα και τις οικονομίες των χωρών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς επειδή είναι πολύ ακριβώς. Και γενικότερα την οικονομία πλήττει κυρίως τις εξαγωγές. Τρίτον, έχουμε διακριτική πρόσβαση στις πρώτες ύλε για την ενέργεια. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται κατά 57% για το φυσικό αέριο, 83% για το πετρέλαιο, 94% για το ουράνιο και περίπου 80% για τον άνθρακα. Ενώ έχουμε δεσμευτεί για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ώστε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, όμως μέχρι το 2040 θα έχουμε κατά 70% εξάρτηση ως Ευρώπη από ενεργειακούς πόρους στενών καυσίμων. Κάτι το οποίο πειράζει πάρα πολύ βέβαια την μακροοικονομική κατάσταση, όπως επίσης και την ανάγκη μας σε επενδύσεις. Θα έπρεπε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και όλα τα αποθεματά τους για επενδύσεις στις υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην διασύνδεση βορρά-νότου, Ανατολής και Δύση. Και γιατί το υπογραμμίζω αυτό. Γιατί πριν μιλούσαμε με τους Πορτογάλους συναδέρφους για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και είναι αλήθεια ότι το ποσοστό που έχουμε πετύχει είναι 70%. Τι έγινε όμως το Δεκέμβριο που μας πέρασε, 18 Δεκεμβρίου, εξαιτία προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την ικανότητα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Βέλγιο και στη Γαλλία, η τιμή στην Ευρώπη έφτασε στα 500 ευρώ ε, στην ε, Χαβατόρα. Εξαιτίας ακριβώς της έλλειψης διασύνδεσης. Τα σύνορα ανάμεσα στη Γερμανία και την Αυστρία. Εκεί διαπιστώσαμε πολύ σημαντική μείωση της συχνότητας και της τάσης στη, στα ηλεκτρικά δίκτυα. Κάτι το οποίο επηρέασε βέβαια την ικανότητα παραγωγής. Είναι σαφές λοιπόν ότι η ανταγωνιστικότητα υποφέρει από αυτή την κατάσταση, ότι οι τιμές υποφέρουν. Υπάρχει αύξηση τιμών που οδηγεί σε καταναλωτές που είναι πιο ευάλωτοι έτσι. Έπειτα υπάρχει διάκριση ανάμεσα στη μία χώρα και στην άλλη, ακόμα και σε περιπτώσεις που θα μπορούσε να υπάρχει δυνατότητα σημαντικής παραγωγής. Υπάρχουν και χώρες οι οποίες υπογράφουν διμερώς συμβάσεις με την Ρωσία. Κάτι το οποίο διπλασιάζει την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελικά από το φυσικό ε, αέριο από 60 δισεκατομμύρια σε 120 δισεκατομμύρια, κάτι το οποίο πλήττει τι οικονομίε πολλών χωρών. Πώς λοιπόν να μιλήσουμε για συνοχή και σύγκληση. Εμείς λοιπόν ως εθνικοί ή βουλευτές ή ευρωβουλευτέ πρέπει να επιβάλλουμε μία τάξη προτεραιοτήτων και έναν χάρτη πορείας για να ολοκληρωθούν αυτές οι επενδύσεις και για να έχουμε επενδύσεις σε εθνικό επίπεδο, για να έχουμε επενδύσεις με επιπτώσεις στις τιμές, που θα επηρεάζουν τις τιμές, και την ικανότητα παραγωγής. Η Πορτογαλία ε, μπλοκάρεται εξαιτία τη διασύνθεση Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία. Ενώ η τεχνολογία μπορεί να μα βοηθήσει σε αυτό, δεν το κάνουμε γιατί θα αυξάνονταν οι τιμέ στη Γαλλία. Θα ήταν όμω υπέρ τη Πορτογαλία. Έπειτα, κάτω χώρε είναι απομονωμένε, δεν υπάρχει διασύνδεση ακόμα. Α σκεφτούμε όμως τα πλεονεκτήματα για την οικονομία των κάτω χωρών, αν υπάρχει αυτή η διασύνθεση. Έχουμε 24 θερματικούς σταθμού. και μόνο το 30% χρησιμοποιούνται. Να λοιπόν, ποια είναι η πρότασή μου. Ελπίζω όλοι να την ακούσουν και να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο τελευταίος θα πάρει το λόγο είναι ο Χάρη Κιάσκαρη, που είναι βουλευτής στο Φιλανδικό Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Uh, thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες ε, και κύριοι. Νομίζω πως οι νέες τεχνολογίες ε, μπορεί να αποτελέσουν απειλή, πρόκληση ή ευκαιρία. Και τις μέρες αυτές ε, κυρίως ασχοληθήκαμε με τις προκλήσεις παρά με τις δυνατότητες. Μιλήσαμε πολύ για την κυρίαση του πληθυσμού δεν συζητήσαμε, παραδείγματος χάρη, πώς ε, το αντιμετωπίζει η Ιαπωνία αυτό με την ε, σύγχρονη τεχνολογία. Μιλάμε συχνά για την εκπαίδευση ότι 40% του πληθυσμού στην Ευρώπη δεν έχει τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Πώς θα αλλάξουμε την εκπαίδευση των δασκάλων λοιπόν για να αλλάξει αυτό. Και μετά σκεφτόμαστε ε, το ότι οι τελευταίε τεχνολογίε έχουν αρνητικά αποτελέσματα στις θέσει εργασία ότι πρέπει να προστατεύσουμε του εργαζόμενου. Πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και επίσης είχαμε μία συζήτηση για το ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας φόρος για τις παγκόσμιες γιγάντιες εταιρείε του διαδικτύου. Πώς θα πρέπει να έχουμε μία πλατφόρμα οικονομιών για να έχουμε και ευρωπαϊκές τέτοιες εταιρείε. Λοιπόν, θα πρέπει άρα να σκεφτούμε διαφορετικά. Εάν ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε την υφιστάμενη τεχνολογία, η κοινωνία θα είναι πολύ διαφορετική. Αν αποφασίζαμε εδώ πέρα στην Ευρώπη να είμαστε πρωτοπόροι. στο να προσαρμοστούμε στην νέα τεχνολογία. Παραδείγματο χάρη στο Κοινοβούλιο της ε, Φιλανδίας συντάξαμε μια έκθεση με τις 11 πιο ριζοσπαστικές τεχνολογίες που επηρεάζουν την ε, κοινωνία μας. Τα αυτόνομα αυτοκίνητα, παραδείγματο χάρη, τα βιομηχανικά ρομπότ, η καθαρή ενέργεια, η οικονομία των ψηφιακών πλατφορμών. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πώς μπορούν αυτά να έχουν θετικό αποτέλεσμα στην ε, κοινωνία μας. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Μια, ένα φιλανδικό εργοστάσιο αυτοκινήτων πριν από 4 χρόνια είχε 800 υπαλλήλους περίπου. Μετά αποφάσισαν ότι θα γίνουν οι πρώτοι στην τεχνολογία της παραγωγής. Παραδείγματος χάρη εγκατέστησαν 600 ρομπότ. Τώρα έχουν 2.500 υπαλλήλους. Οπότε η δημιουργία της τελευταίας τεχνολογίας μπορεί να σημαίνει και περισσότερες θέσεις εργασίας, όχι το αντίθετο και μετά γνωρίζουμε ότι γύρω στο 15% του τζίρου γίνεται σε ψηφιακές πλατφόρμες Amazon, Google, Alipay αλλά σε 15 χρόνια θα είναι γύρω στο 50% στις πλατφόρμες αυτές οπότε πρέπει να το σκεφτούμε αυτό θα πρέπει να έχουμε μήπως ευρωπαϊκές ψηφιακές πλατφόρμες και εταιρείε αντί να προσπαθούμε να φορολογούμε τις εταιρείε των άλλων. Μετά. Σημειώνω ότι πρέπει να μειώσουμε και τις εκπομπές μας ε, από τις μεταφορές ε, κατά 5% μέχρι το 2030. Στην ε, Φιλανδία Κάναμε μια υποχρεωτική κατανομή, δηλαδή 30% όλων των καυσίμων θα πρέπει να είναι βιοκαύσιμα. Τώρα έχουμε μία από τις ε, κορυφαίες εταιρείε στον κόσμο που παράγει βιοκαύσιμα στη Φιλανδία, ε, λόγω αυτού του κανονισμού. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δυνατότητες επίσης της κυκλικής οικονομίας γνωρίζουμε τώρα ότι χρησιμοποιούμε τα υλικά άπαξ. Πάνω από 30% των τροφίμων πετάγεται. Και χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητά μας μόλις 8% του χρόνου. Πώς ε, θα έπρεπε να έχουμε κάποιες ευρωπαϊκές εταιρείες που να ασχολούνται με αυτά. Και τέλος. Υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ε, ήδη τώρα ένα σύστημα εντελώς καθαρής ενέργειας. Ήδη στη Φιλανδία 80% της παραγωγής ενέργειας είναι χωρίς ε, διοξείδιο του άνθρακα και τώρα δημιουργούμε ένα έξυπνο σύστημα ενέργειας ε, που αφορά την αποθήκευση, το ευέλικτο που θα μπορούσε ακριβώς ε, να μας πάει σε μια νέα καινοτόμο σκέψη οικοσύστημα το λέμε. Βλέπετε λοιπόν ότι στηρίζουμε τα προγράμματα αυτά Invest EU, υποστηρίζουμε την καινοτομία και την πολιτική που βασίζεται στην καινοτομία και το φθινόπωρο όταν θα αναλάβουμε την ε, Προεδρία σας περιμένουμε στο Ελσίνκι για να κάνουμε κάποια καινούργια πράγματα μαζί. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή. Και τώρα θα δώσω το λόγο σε εσά που ζητήσατε να παρέμβετε σε αυτή τη συζήτηση. Ο πρώτος θα είναι ο κύριος Ανδρέα Μπερκέγκερ από την Bundestag, Γερμανία. Ja, ε, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω λίγα λόγια. Το πρόγραμμα InvestEU είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς ε, μπορεί να παίξει θετικό ρόλο η κρατική παρέμβαση στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης ε, θετικό παράδειγμα για το πώς ε, μπορεί να υπάρξει η συνεργασία των κατοικοφορέων για να βελτιωθεί η λειτουργία τους. Ε, είδα την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και βλέπουμε ότι αξιολογήθηκε ένα από τα προγράμματα που προηγήθηκε του ΕΦΣΥ και εάν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε τα συμπεράσματα αυτά για το ΕΦΣΥ νομίζω έχουμε ένα καλό παράδειγμα του πώς μπορούμε να βελτιωθούμε. Ακούστηκαν πολλά για αυτό το θέμα. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στον κύριο Χόιερ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων, που σωστά είπε ότι δεν μπορούν αυτές οι επενδύσεις να γίνουν μόνο με δημόσια χρήματα. Πρέπει να υπάρξει και ιδιωτική χρηματοδότηση, γιατί είναι περιορισμένα τα κρατικά κονδύλια. Γι' αυτό εγώ θεωρώ, εμεί θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αυτό Πρέπει βεβαίως ε, να το υποδεχτούμε θετικά, ειδικά δεδομένων των εξελίξεων των επομένων ετών, το κενό του, της χρηματοδότησης που θα προκύψει από το Brexit και τις νέες δαπάνες ε, λόγω των νέων ε, αρμοδιοτήτων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε χαιρετίζουμε το ότι έχουμε μέχρι και 14 μέσα τα οποία ενώνονται εδώ πέρα. Έχουμε διάφορα πλέον εκτήματα θα αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη και αν έχω καταλάβει σωστά θα μπορέσει να ανέβει και η σχετική αξιολόγηση οπότε ε, θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το σύστημα απρόσκοπτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε κάποιες επιφυλάξεις αλλά η μόχλευση η οποία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή και μας ε, έπεισε. Βλέπουμε ότι είχαμε μέχρι 650 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία μπορούν να προκύψουν ως επενδύσεις. Έχουμε δηλαδή κάτι το οποίο θα μπορέσει να καλύψει ένα μεγάλο μέρος του κενού των επενδύσεων που δεν μπορεί να καλύψει η αγορά. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρχει πολιτική στόχευση για την ενίσχυση της καινοτομίας ε, των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των κοινωνικών επενδύσεων και οπωσδήποτε της ε, αηφόρου υποδομής ένα μήνυμα που πρέπει να στείλουμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί και στο μέλλον απέναντι στις ΗΠΑ και άλλες χώρες όπως η Κίνα. Οπότε δεν μπορώ παρά να στηρίξω αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Μανουέλ Καλδέρα Καμπράλ. Από την Εθνοσυνέλευση της Πορτογαλίας. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω αυτήν την πρωτοβουλία, ένα πολύ σημαντικό βήμα για να προωθήσει τις επενδύσεις και την καινοτομία και την συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και την επένδυση στην αηφορία. Είναι ενδιαφέρον νομίζω το ότι έχουμε μια εγγύηση του 75% και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το υπόλοιπο 25% που ε, θα καλυφθεί από τα κράτη-μέλη να δούμε πώς ε, θα ελέγχεται από πλευράς ε, δημοσίων λογιστικών επίσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και τα εθνικά διαρθρωτικά κονδύλια αλλά να δούμε και τους περιορισμούς που έχουν καμιά φορά αυτά τα ταμεία ε, που σημαίνει λιγότερη ευελιξία. Μία τέταρτη ιδέα που θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι επίσης το ότι τα μέσα αυτά θα πρέπει να είναι πιστώσεις αλλά και με μετοχικό κεφάλαιο και επενδύσεις ειδικά για να προωθήσουμε την ε, καινοτομία, τις νέες επιχειρήσεις ε, και την ψηφιακή επανάσταση. Η τελευταία ιδέα είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα ταμεία αυτά να επιτρέπουν την επένδυση στον τομέα της ψηφιοποίησης όχι μόνο για τις εταιρείε, αλλά και στις υποδομές όπου θα έχουμε σημαντικές ε, προκλήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει τώρα ο Κύπριος ε, συνάδελφός μας, ο κύριος Μαυρίδης, Ευρωβουλευτής. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι επενδύσεις είναι κινητήριος μοχλός της βιώσιμης ανάπτυξης, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, της κοινωνικής πρόοδου και της ευημερία. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε την προβλεπόμενη αύξηση των κοντιλίων του προγράμματος Ορίζοντας 2020 για έρευνα και καινοτομία στο πλαίσιο του νέου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, καθώ και την προβλεπόμενη αύξηση τη χρηματοδότηση για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, γεγονό που εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Η Κύπρος έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η έλλειψη χρηματοδοτήσεων και στενότητα επενδύσεων συνεπία της απόφασης της Ευρωομάδας για απομείωση καταθέσεων, το γνωστο Μπέιλιν, τον Μάρτιο του 2013, γονάτισε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας. Επίσης, ο δυσανάλογα προς τον πληθυσμό της, μεγα... της μεγάλος αριθμός παράνομων μεταναστών ή αιτητών ασύλου που δέχτηκε η Κύπρος έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε σε σχέση με τη διασφάλιση χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης και την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία παραμένουν στην κυπριακή οικονομία αποτελώντας το 31% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Είναι εδώ που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει έμπρακτη αλληλεγγύη προς την Κύπρο μέσω της προώθησης τη ανάπτυξη και των επενδύσεων στη χώρα μα, αλλά και τη ισότιμη κατανομή βαρών σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Η Κύπρο, παρά τη στενότητα επενδύσεων, δεν επωφελήθηκε ιδιαίτερα από το επενδυτικό σχέδιο Juncker. Προσβλέπουμε ότι το νέο επενδυτικό σχέδιο InvestEU θα είναι πιο φιλικό και προσβάσιμο, ώστε να παρέχεται ισότιμη δυνατότητα και σε μικρέ χώρε όπω η Κύπρο για απορρόφηση κονδυλίων. Εκτιμούμε ότι η Κύπρος θα μπορούσε να αξιοποιήσει το πρόγραμμα InvestEU για ανάπτυξη των ακόλουθων τομέων των ενεργειακών υποδομών, ιδιαίτερα εν ώψη τη εξόριξη φυσικού αερίου, τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και τη έρευνα και καινοτομία. Καταλήγοντα, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη τα χρηματοδοτικά εργαλεία τη ΕΕ να συνεχτιμούν τι ιδιαιτερότητε που παρουσιάζει το κάθε κράτο μέλο τη Ένωση χωριστά παρέχοντα πρόσθετα χρηματοδοτικά κίνητρα, παραδείγματο χάρη η Κύπρο είναι απομονωμένη αγορά μικρού μεγέθου, χωρί χερσαία διασύνδεση, με αποτέλεσμα να διαθέτει περιορισμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Σα ευχαριστώ και επί την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Προεδρείο και όλου του διοργανωτέ για τη φιλοξενία, όπω επίση και του αγαπητού μεταφραστέ, που σίγουρα είναι οι μόνοι που έχουν ακούσει με προσοχή όλε τι ομιλίε. Merci. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μοσκουστάροβιτς, Σλοβενία. Από το Σλοβενικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ κύριε Στάροβιτς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήδη για το 2020 ξέρουμε ότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις δίνουν αποτελέσματα και οι επενδύσεις αυτές πρέπει να αποτελέσουν μέρος και των επενδύσεων στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021 2027. Γι' αυτό λοιπόν εγώ συστήνω μέρος των επενδύσεων αυτών να πάνε και σε κοινωνικά προγράμματα. Πρέπει να έχουμε λύσεις πιο αποτελεσματικές προκειμένου να σταθεροποιηθεί ο δημόσιος τομέας. Είμαι πεπισμένος ότι η γνώση μπορεί να μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε καλές πολιτικές, ακολουθώντας το πνεύμα του Αριστοτέλη, για τον οποίο η πολιτική είναι μια δραστηριότητα ελεύθερων ανθρώπων για να πετύχουν μια δίκαια και συντεταγμένη κοινωνία. Τέλος, θα ήταν πολύ χρήσιμο να ερευνήσουμε περισσότερο τι γίνεται με το ΣΕΡΝ, το ερευνητικό αυτό κέντρο. Σίγουρα μπορεί να μας δώσει πολλές πληροφορίες που θα ήταν χρήσιμες ε, για μας για να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε σε μια κοινωνία όλο πιο περίπλοκη και ασταθής. Οι λύσεις δεν είναι απλές. Απλές ε, λύσεις προτείνουν μόνο οι λεκιστές. Σήμερα βλέπουμε ότι τα δεδομένα είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Τα big data είναι πολύ χρήσιμα αλλά χρησιμοποιούνται πολλές φορές περισσότερο για τη χειραγώγηση παρά για το καλό της κοινωνίας. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τη γνώση και τους μηχανισμούς αυτούς ώστε να βελτιώσουμε την κοινωνία και να προσανατολιστεί ώστε να τηρήσει τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης και τον κοινωνικό πυλώνα της Ευρώπης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Μαργαρίτα Μάρκες, που είναι από το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Ehm, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο για τις παρουσιάσεις τους, τον ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ελεκτικού Συνεδρίου. Μιλάμε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Περιορίζονται τα ποσά ε, συνοχής από την Επιτροπή τα επιμερισμένα κονδύλια και αυξάνονται αυτά που έχουν να κάνουν με την άμεση διαχείριση. Όμως ακριβώς αυτά τα τελευταία είναι που πρέπει να περιλαμβάνουν μια μεγάλη συνιστόσα συνοχή. Στον προπολογισμό αυτό λοιπόν έχουμε και το πρόγραμμα Invest EU. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν θα πρέπει να συγκεντρώνει πολλά στοιχεία πολλούς μηχανισμούς και τους εσωτερικούς, γιατί το πρόγραμμα αυτό μας επιτρέπει να εξορθολογήσουμε, να κατανοήσουμε καλύτερα και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Αν κατευθύνεται στην τεχνολογία, στην καινοτομία, την ε, κλιματική αλλαγή, τη βιομηχανία κλπ, δεν πρόκειται για μια οποιαδήποτε επένδυση. Θα πρέπει να πρόκειται για επενδύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το μέλλον και άρα με τις προτεραιότητές μας. Και θα πρέπει οι επενδύσεις αυτές να ενισχύουν τη συνοχή. Και για να προωθηθεί συνοχή είναι αναγκαίο το πρόγραμμα αυτό να διαθέτει κανόνες ώστε να τηρείται και η γεωγραφική κατανομή, η ισορροπία δηλαδή στη γεωγραφική κατανομή. Είναι πολύ σημαντικό που ακούσαμε την εκπρόσωπο του λεκτικού συνεδρίου που αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Juncker και μας είπε ότι από τη στιγμή που υπήρξε τροποποίηση στον κανονισμό για να προωθηθεί η γεωγραφική ισορροπία, η ισορροπία αυτή έγινε πραγματικότητα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το Invest EU και αυτό το πρόγραμμα να προωθήσει την γεωγραφική ισορροπία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο και πάλι στον κύριο Κώστα Μαυρίδη, γιατί πριν όταν ε, τον ε, κάλεσα, είναι ο ευρωβουλευτής μας που εκλέγεται στην ε, Κύπρο, τελικά ήταν ο κύριος Βόρτσης που πήρε το λόγο. Οπότε, ο κύριος Μαυρίδης τώρα. Vous Is working? Yes, it is. I my mother tongue. Θα είμαι σχετικά σύντομος. Νομίζω ότι έχουν λεχθεί πάρα πολλά σωστά πράγματα γύρω από τον ευρύτερο στόχο για να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με πραγματική σύγκληση των οικονομιών και των κοινωνιών μας, όπως ήταν και το αρχικό όραμα των δημιουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτων λεχθέντων όμω, θα ήθελα να πάρω τη συζήτηση σε δύο πολύ συγκεκριμένα θέματα, που συζητάμε πάρα πολύ έντονα και στην Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρώτο είναι ότι συγκεκριμένα κράτη-μέλη έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση με ένα πολύ βάναυσο τρόπο και ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης αποφασίστηκε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα από αυτά που αποφασίστηκε είναι το πλαίσιο η αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης με τρεις πυλώνες κοινούς κανόνες εποπτείας, κοινούς κανόνες επίλυσης προβληματικών τραπεζών και πανευρωπαϊκό σχέδιο εγγύησης καταθέσεων. Σας μιλώ σαν οικονομολόγος. Δεν αποδέχομαι τα πολιτικά επιχειρήματα που προβάλλονται σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρεμποδίζεται η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης με πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων. Κατανοώ ότι υπάρχουν προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά αυτό δεν είναι αιτιολόγηση για την καθυστερούμενη κατάσταση που βλέπουμε. Και θα το θυμηθούμε αυτό μπροστά στην επόμενη τραπεζική κρίση. Τότε κάποιοι από εδώ θα ζητούν συγγνώμη, αλλά θα είναι αργά. Το δεύτερο, και τελειώνω, είναι ότι η εμπειρία μου ως εισηγητής στο πρόγραμμα, για, για, στο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για τις υποδομές μπορώ να πω ότι ήταν πολύ επιτυχημένο βλέποντας και ποιοι επωφελήθηκαν από το γεγονός ότι δώσαμε ιδιοκτησία, το ownership, το δώσαμε πίσω στα κράτη-μέλη. Όχι δια της επιβολής, αλλά μέσα από τον δικό του σχεδιασμό. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θα μείνω μόνο σε αυτά τα δύο γιατί θέλω και αυτά να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Αλής Μαργίγκινς που είναι γερουσιάστρια από την Ιρλανδία. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς επενδύσεων. Το γνωρίζω ως ε, Ιρλανδοί καθώς αντιμετωπίζουμε την μετάβαση στην κατάσταση του Brexit ε, και την επίγουσα μετάβαση που απαιτείται σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Αλλά για να απαντήσω σε κάποια από αυτά τα οποία ακούστηκαν σε σχέση με την ε, κλιματική αλλαγή και τους στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ βεβαίως έχει σημαντικό ρόλο να παίξει ο ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να γίνουν οι στόχοι αυτοί κερδοφόροι. Γι' αυτό πρέπει να λάβει έναν ρόλο ο δημόσιο τομέα. Γι' αυτό οι επενδύσει ή οι δημόσιε για να υπάρξει αυτή να αντιμετωπιστεί αυτή η μείωση κατά 20% των δημοσίων επενδύσεων πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα γιατί και ο δημόσιος είναι σε θέση να κινητοποιήσει την καινοτομία και στην εφαρμοσμένη και στην βασική έρευνα και βεβαίως ε, να προχωρήσει σε κινήσεις ε, μεγάλης ε, κλίμακας και βεβαίως να προχωρήσουμε και σε μεταφορές προς τον παγκόσμιο νότο. Λοιπόν, χάρηκα επίσης για το ότι μιλάμε για την ευελιξία όσον αφορά το ότι κάποιοι κανόνες ε, περί δημοσίων επενδύσεων καμιά φορά έχουν ε, ένα αποτέλεσμα αρνητικό στο πώς αντιμετωπίζεται ακριβώς ε, οι επενδύσεις όσον αφορά τα συστήματα επενδυτικών δικαστηρίων στις πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες και βεβαίως η ρήτρα αυτή μη υπαναχώρησης που ακριβώς καθιστά δύσκολο να πάμε από μια ιδιωτική σε μια δημόσια παροχή υπηρεσιών εκεί όπου μπορεί να γίνει αυτό. Πρέπει λοιπόν να δούμε τις διαπραγματευτικές έντολες στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες για αυτό το θέμα. Τέλος, παρατηρώ ότι υπάρχει μια αύξηση από 2,2 εκατομμύρια στα ε, δισεκατομμύρια στα 4 δισεκατομμύρια όσον αφορά τις κοινωνικές επενδύσεις αλλά είναι ακόμη πολύ χαμηλότερο από τα 11 δισεκατομμύρια τα οποία επενδύονται στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη αηφόρου βεβαίω υποδομή, την οποία υποστηρίζω, αλλά σε ζητήματα όπω η φροντίδα του πληθυσμού, ο οποίο και κάτι το οποίο αναφέρθηκε. Ζητήματα όπω η αναπτύξη των κοινοτήτων, υποδομέ ισότητα. Αυτά είναι κοινωνικέ υποδομές και αναρωτιέμαι όλα αυτά θα πάνε από τι κοινωνικέ επενδύσει ή μπορούμε να, επενδύσουμε, επεκτείνουμε αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε ως ε, επενδύσεις στις υποδομές, ειδικά μετά από μια περίοδο στην οποία έχουν ατροφήσει. Και βεβαίως, όπως είπαμε, η φροντίδα είναι ο τομέας έντασης εργασίας του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ο Ιγκόρ Πιμένοφ από την Λιθουανία. Τη Λετωνία, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα προς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον κύριο Βέρνερ Χόιερ, αλλά βλέπω ότι έχει φύγει. Παρ' όλα αυτά, θα απευθύνω την ερώτησή μου στα υπόλοιπα μέλη του πάνελ. Ο κύριος Χόιερ είπε ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στις ε, δημόσιες επενδύσεις και πρέπει να κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Ε, δεν είναι ακριβώς η δημόσια ε, επενδυτική ε, και αναπτυξιακή τράπεζα κάτι ανάλογο με την KfW της ε, Γερμανίας. Η κατάσταση στην χώρα μου, γενικά μιλώντας, είναι σαν την Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Οι Γερμανοί επιχειρηματίες δεν είχαν καθόλου λεφτά τότε, καθόλου ασφάλεια και λίγοι άνθρωποι σε ηλικία εργασία. είχαν μείνει και στην ε, δική μου τη χώρα έφυγαν πάρα πολλοί νεαροί άνδρες για τι δυτικέ ε, χώρε τη Ευρωπαϊκής Ένωση για να βρουν δουλειά και η βιομηχανία έχει περιορίσει την παραγωγή της στο 1 τρίτο της παραγωγής του 1989. Η Γερμανία το έλυσε αυτό με την σύσταση μιας σειράς τραπεζών που ανήκαν στην Ομοσπονδιακή και κυβέρνηση και στα τοπικά κρατήρια που επένδυσαν και έτσι είχαμε ανάπτυξη και δουλειά στο γερμανικό σύστημα που δείχθηκε πολύ επιτυχημένο και διασφάλισε το μεταπολεμικό οικονομικό θαύμα και τώρα είναι η πιο επιτυχημένη χώρα στην Ευρωζώνη. Οπότε το εάν οι δημόσιες αναπτυξιακές ε, τράπεζες είναι εντός των επενδυτικών ε, προτεραιοτήτων για την περίοδο μετά το 2020. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Λίβ Βίρινγκς, Ευρωβουλευτής. Ε, σας ευχαριστώ. Δεν έχω όμως ε, ερωτήσεις. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ah bon. Χρησιμοποίησατε το χρόνο σα, σας δηλαδή. Ωραία. Τελευταίος που θα πάρει το λόγο, η κυρία Γκαμπρίελα Κρετού από την Γερουσία της Ρουμανίας. Γερουσιαστής λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν μπορώ παρά να σας υπενθυμίσω ένα σχόλιο που έκανα νωρίτερα πέρυσι στη διάσκεψή μας για το σχέδιο Juncker που εισήχθη μια νέα ιδέα. Υπάρχουν κακές επενδύσεις, άμεσες δημόσιες επενδύσεις που πρέπει να αποφεύγονται γιατί υπονομεύουν την δημοσιονομική σταθερότητα και υπάρχουν και ιδιωτικές που χρησιμοποιούν όμως ως κίνητρο δημόσιο χρήμα σαν εγγύηση. Όλα αυτά είναι ιδεολογίες όμως, δεν είναι οικονομική πολιτική. Η ιδεολογία από μόνη της Τίποτα το κακό. Αλλά όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ήταν επιτυχία το σχέδιο Juncker, αλλά η περίοδος είναι τόσο σύντομη που είναι δύσκολο να το πούμε και να πούμε σε τι βαθμό εξαρτηθήκαμε ε, στην ιδιωτική πίστη και τι θα γίνει αν ακολουθήσουμε τη ίδια στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ νωρί για να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση και να ξέρουμε ε, τι όφελος προσφέρει αυτού του είδους η επένδυση στο κοινό όταν βασίζεται μόνο σε χρηματοδοτικά μέσα. Εγώ πιστεύω, όπως είπα και νωρίτερα, ότι πρέπει να εφεύρουμε ε, αγαθά, υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, σημερινή κοινωνική δυσαρέσκεια που εκφράζεται από τις κοινωνίες μας. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, καλώς. Όσοι ήθελαν να πάρουν το λόγο, μίλησαν. Μας μένει λίγος χρόνος ακόμα, οπότε θα δώσω το λόγο τώρα στους ε, υπόλοιπους για να τους ζητήσω να πάρουν το λόγο αν θέλουν ε, δεδομένων των παρατηρήσεων που έγιναν. Η κυρία Τερτόπνου πρώτα απ' όλα από το Ελεκτικό Συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Για το ερώτημα του πόσο σημαντικό είναι ο ιδιωτικό τομέα και οι ιδιωτικέ τράπεζε βεβαίω είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί όπω ξέρετε για το FC και το επισημάναμε αυτό και στην ε, δεύτερη απάντησή μας ότι θα πρέπει το FC να προσπαθήσει να αποφύγει τον ανταγωνισμό με άλλες πηγές ε, κοινοτικής ε, χρηματοδότησης αλλά και με τον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω πως η δύναμη ακριβώ της συνεργασίας στο InvestEU EU είναι το ότι μπορεί να υπάρχει ένα αποτέλεσμα πολλαπλασιαστικό και να ενισχυθούν και οι δύο πλευρές. Αυτή είναι η απάντησή μου. Και νομίζω ότι θα ζητούσα και από τους συναδέλφους εδώ πέρα να δουν την έκθεσή μας, ειδικά την δεύτερη σύστασή μας και την δεύτερη πρόκληση που αναφέρουμε εκεί. Σας ευχαριστώ. Χωσέ o InvestEU. Σας ευχαριστώ. Το InvestEU βεβαίω είναι και δημόσιε και ιδιωτικέ επενδύσει. και ελπίζω έτσι ότι θα μπορέσουμε να κλείσουμε ένα κενό του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του ΕΦΣΥ, γιατί χρειαζόμαστε υποδομές και διασυνοριακές πλατφόρμες επενδύσεων στις οποίες θα συμμετέχουν και τρίτες χώρες έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να προσφέρει αυτήν την ε, εγγύηση και εδώ πέρα συμφωνώ μαζί σας όσον αφορά τις ε, διασυνδέσεις. Αυτό υπάρχει σε όλα τα προγράμματα και στο InvestEU αλλά μπορούμε να έχουμε μια ενεργειακή ένωση, μια ψηφιακή ένωση αν ταυτόχρονα υπάρξουν αυτές οι συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων χωρών και το ΕΦΣΙ είχε ήδη ένα τέτοιο κομμάτι αλλά εδώ πέρα θα πρέπει να παραμερίσουμε τα όρια που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων μονάδων. Μετά, για την κλιματική αλλαγή, να σας υπενθυμίσω εδώ ότι 40% των επενδύσεων είναι δεσμευμένες ακριβώς για την ε, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μεταξύ του 2021 και 2025 ε, θα αυξηθούν και από το 2027 θα πρέπει κάθε χρόνο να επιτυχάνουμε το 30%. Τα, τα κοινωνικά ζητήματα είναι σαφές ότι το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ασχολείται και με τα θέματα τα κοινωνικά αλλά μόνο 4% του υφιστάμενου σχεδίου έχει οριστεί για τα κοινωνικά. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται βεβαίως μια ενίσχυση και έχουμε ακριβώς να στηρίξουμε όλους αυτούς τους οργανισμούς κοινωνικής αλληλεγγύης και προσπαθούμε ακριβώς να κινητοποιήσουμε άλλα επιπρόσθετα 95 εκατομμύρια ευρώ ε, για τον ε, τομέα αυτό. Βλέπουμε όμως ότι δεν εξαντλούνται τα ποσά γιατί δεν επαρκεί η ζήτηση. Όσον αφορά τις ε, συνεισφορές θα ήθελα να υπενθυμίσω πως έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εκτός του ΕΦΣΥ e, μάλιστα υποστηρίζουμε την ε, οικονομία. Υπάρχουν 79 δισεκατομμύρια ευρώ που πρέπει να τα αναφέρουμε. Και τέλος μια παρατήρηση. Υπάρχει και το θέμα της επιχειρηματικότητας που πρέπει να ενισχύσουμε και μέσω ακριβώς του μετοχικού κεφαλαίου το κάνουμε και αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Φερναντές γιατί υποκαταστήσατε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο κύριος Γιάνκο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που προσφέρουν λύσεις στις ε, υφιστάμενες προκλήσεις και που τα ξεχάσαμε. Υπάρχουν στα επενδυτικά σχέδια. Μιλήσαμε, ξεχάσαμε να μιλήσουμε για την ευαλωτότητα της αγοράς εργασίας και για τους ανθρωπίνους πόρους και το κεκτημένο που αποτελούν οι ανθρώπινοι πόροι σε όλη την Ευρώπη σε ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο είναι ολοένα και πιο εχθρικό, σε ένα γεωπολιτικό πλαίσιο το οποίο είναι ολοένα και πιο εύθραυστο και ευαίσθητο ε, σε διάφορες περιφέρειες. Η πρόσβαση της Ευρώπης στις πρώτες ύλες, η διατήρηση της Ευρώπης ως μιας ποιοτικής αγοράς, εξαγοράς, εξαγωγής τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, η παρουσία της Ευρώπης με προστιθέμενη προστιθέμενη αξία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις ε, αϊφόρες τεχνολογίες. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε εξοπλισμό που μας βοηθά να καταπολεμήσουμε τις παρενέργειες και τις δυσάρεστες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά και πρέπει να τα συντονίσουμε καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε πρόσβαση όλων των χωρών, αυτό πρέπει να έχουμε, με μη διακρισιακό τρόπο, χωρίς διακρίσεις, σε αυτό Το που αποτελεί το πιο σημαντικό κόστος σε οποιαδήποτε παραγωγή, που είναι το κόστος ενέργειας για να τροφοδοτηθεί ενέργεια που θα δημιουργήσει αυτή την παραγωγή. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν πέσει σε αυτό το φαύλο κύκλο, διότι οι πολιτικές για τους διαδρόμους τους ενεργειακούς το μόνο που κάνουν είναι να απομακρύνουν κάποιες χώρες. Οι αγωγοί δεν παίρνουν από αυτές τις χώρες, οι οποίες φτωχαίνουν και άρα έχουμε μαζική μετανάστευση ε, του εργασιακού δυναμικού από τις χώρες αυτές. Δεν καταλαβαίνω και δεν μπορώ να κατανοήσω πώς κανείς καταρτίζει ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ε, χωρίς να κάνει διακρίσεις. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο εγχείρημα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ναι, αν υπήρχαν μικρότερες αποκλήσεις στην τιμή της ενέργειας, οι μισθοί θα αυξάνονταν γρηγορότερα στη Ρουμανία. Σας ερωτώ. Εξαιρετικό το ερώτημά σας, κύριε Πρόεδρε. Αν δούμε Σύνεγγι στα ευρωπαϊκά έργα αναφορικά με τους διαδρόμους μεταφοράς των υδρογονανθράκων προς την Ευρώπη, τότε θα παρατηρήσουμε ότι όλοι αυτοί οι αγωγοί δεν περνούν από τη Ρουμανία και έτσι η Ρουμανία γίνεται εχμάλωτη της Ρωσίας, Όμηρος, η οποία διατηρεί πολύ υψηλές τιμές στην προμήθεια φυσικού αερίου για τον ενεργειακό ανεφοδιασμό. Τα ρουμανικά προϊόντα πλήττονται και η ανταγωνιστικότητά τους μειώνεται τα μάλα. Επομένως, θεωρούμε ότι ένας μεγάλος ε, ε, ε, Οικονομικό παίκτη Ευρωπαίος στην Ρουμανία, κλείνει τα εργοστάσια στη Ρουμανία και επιστρέφει στη χώρα του. Με όλα αυτά τα δυσάρεστα, με αυτές τις δυσάρεστες εξελίξεις έχουμε ρουμανικό εργασιακό δυναμικό που μεταναστεύει προς τις χώρες μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση τη ρουμανικής οικονομία. Ευχαριστώ. Φτάνουμε στο τέλος αυτής της ανταλλαγής απόψεων, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, πλούσια και πολλά υποσχόμενη. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που παρέστησαν εδώ, στο πάνελ που ε, ήταν από την αρχή της συνεδρίασής μας και έκαναν παρουσιάσεις. Δίνω το λόγο στον Σορίν Λαζάρ, ο οποίος συμπροέδρευσε για τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προτιμήσω να μιλήσω ρουμανικά, επιτρέψτε μου. Αξιότιμε πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι η βασική πολιτική επενδύσεων είναι η περιφερειακή και η πολιτική συνοχή. Η περιφερειακή πολιτική απευθύνεται σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηρίζει την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, την βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα της ζωής. Η πολιτική συνοχή αποτελεί καταλήτη για επιπλέον χρηματοδότηση και επιβάλλει στις χώρες μέλη συγχρηματοδότηση από το εθνικό επίπεδο και έτσι υπάρχει και περισσότερη εμπιστοσύνη από τους επενδυτές. Η Ρουμανία λοιπόν βλέποντας τις προτεραιότητες για μετά το 2020 ε, θεωρεί ότι μία ισορροπημένη κατανομή και ισόρροπη γεωγραφικά των επενδύσεων αυτών ε, μπορεί να συνεισφέρει στην μείωση των σημαντικών αλλαγών, ε, διαφορών συγγνώμη, στην ανάπτυξη μεταξύ χωρών και περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να συνοψίσω κάπως τα όσα ακούσαμε σήμερα εδώ. άκουσα πολλά και διάφορα θέματα και ερωτήσεις που περιμένουν κάποια λύση, σύντομα κάποια απάντηση. Η διαφορά στην παραγωγικότητα ανάμεσα σε εμά, την Ασία και τις Ηνωμένε Πολιτείε πρώτα απ' όλα, ότι πρέπει να επενδύσουμε στην κοινοτομία, την έρευνα, τι υποδομέ, τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον κοινωνικό τομέα, στι ανανεώσιμε ενέργειες, αλλά και σε άλλου τομεί όπου δεν έχουμε σήμερα ιδιωτικό κεφάλαιο. Επίσης μιλήσαμε για την αναγκαιότητα να κινητοποιήσουμε ε, ιδιωτικά κονδύλια επιπλέον από τα κρατικά. Είπαμε ότι το InvestEU δεν πρέπει να αντικαταστήσει την πολιτική συνοχής, ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία, επενδύσεις σε δημόσιες πολιτικές. Επίσης, Μιλήσαμε και για την παρουσία του ιδιωτικού τομέα που είπαμε ότι πρέπει να κάνει μια παραπάνω προσπάθεια και να συμβάλλει και αυτό στην μείωση της κλιματικής αλλαγής. Μιλήσαμε για την Κεντρική Τράπεζα και είπαμε ότι μπορεί να αποτελέσει μοντέλο αναπτυξιακό. Να λοιπόν σημαντικά θέματα τα οποία περιμένουν μια απάντηση και μάλιστα γρήγορα. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ως βουλευτής και πολίτης της Ρουμανίας αλλά και πολίτης της Ευρώπης επιθυμώ περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη διαφάνεια για την Ρουμανία και περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη ανταγωνιστικότητα, περισσότερη αποτελεσματικότητα και περισσότερη πειθαρχία. Είμαι πεπισμένος ότι και εσείς θέλετε τα ίδια για τις χώρες σας. Αλλά θέλω επίσης και περισσότερη αλληλεγγύη και περισσότερη συνοχή για να υπάρξει μια πραγματική σύγκληση στην Ευρώπη. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνο εφόσον παραμείνουμε ενωμένοι. Μόνο τότε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα και τόσο απρόβλεπτα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρου του Ρουμανικού Κοινοβουλίου χαιρετίζω την παρουσία όλων εδώ στην εκδήλωση αυτή και επαναλαμβάνω την πεποίθησή μου ότι μαζί θα βρούμε τον καλύτερο δρόμο για να χαίρουμε ευημερίας όλοι. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ πολύ όλους. Είχαμε δύο ημέρες με διάφορες συναντήσεις μεταξύ εθνικών βουλευτών και ευρωβουλευτών. Αποτελεί μια σημαντική στιγμή και νομίζω ότι όλοι έχουμε κάθε συμφέρον να βρούμε σημεία συνάντησης μεταξύ μας για να υπάρχει πλήρης κατανόηση για τα όσα γίνονται στα εθνικά κοινοβούλια και τα όσα γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές οι δύο μέρες πρέπει να έχουν συνεισφέρει σε αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχει πρόοδο στο περιεχόμενο των συναντήσεων αυτών, στην ποιότητα των ε, ανταλλαγών που έχουμε μεταξύ μας. Είναι αλήθεια ότι η βούληση για μια αλληλέγγυα Ευρώπη είναι κοινή. Για μια Ευρώπη η οποία ετοιμάζει το μέλλον όλων των Ευρωπαίων. Για μια Ευρώπη επίσης που μας προστατεύει απέναντι στι προκλήσεις που μας στέλνει η παγκοσμιοποίηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και τον καθένα από εσά χωριστά για τη συμμετοχή σας εδώ.